την ε, ευχαρίστηση να σας ανακοινώσω ότι αυτή η συζήτηση περιέχει μόνο δύο ομιλητές. Την κυρία Ίντβελτ και τον κύριο Μπαρνιέ. Και, και περίπου 40 ανθρώπους που έχουν ζητήσει το catch the eye. That's not true. Okay, so, Sophie Ίντβελτ, you have the floor for four minutes. Κυρία Ίντβελτ, έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και οι συνάδελφοι που τώρα φεύγετε Είχαμε πάρα πολύ ευρία πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αυτό είναι καρπός της κοινή προσπάθειας από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου να ευχαριστήσω και τους κοιόδες επόμενου ηγητέ που εδώ πέρα παρίστανται ακόμα γιατί ήταν πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Και επίση μας βοήθησε πάρα πολύ και η προηγούμενη επιτροπή η κυρία Κρόου γιατί ο καταναλωτή ήταν στο επίκεντρο τις, τις πολιτικές του καταναλωτή που θέλουν. Αλλά και ο Επίτροπος Αλμούνια βοήθησε. Οπότε να δούμε τώρα τι έγινε με τα καρτέλ. Γιατί σε σχέση με τα καρτέλ συζητήθηκε πάρα το πως θα έχουμε κάποιε αποτελεσματικές κυρώσεις ε, πρόστιμα, ποινικέ κυρώσει. όμως πριν επισέλθουμε ή στι λεπτομέρειε θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι εταιρείε για να αποφύγουν τις κυρώσεις δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε καρτέλ γιατί νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν τις αρχές του ανταγωνισμού ε, γελιώνται ουσιαστικά το μόνο το οποίο κάνουν είναι να επιβαρύνουν τον καταναλωτή τα καρτέλ μόνο ένοχα είναι, δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε κυρώσει σε τέτοιες συμπεριφορές ιδίως ε, να έχουμε κάποιους οι οποίοι επαναλαμβάνουν το παράπτωμα Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε υπάρχει αναλογικότητα, μην είμαστε υπερβολικοί με τις ε, κυρώσεις και τα πρόστιμα, να μπορούμε να επεξεργαστούμε περισσότερο, να χτενίσουμε αυτά τα μέτρα κυρώσεων και να δούμε κάποια επιμέρους θέματα όπως η ατομική ευθύνη, η διαφάνεια, η λογοδοσία, οι διαδικασίες, η, η η, η δίκαιη δίκη των εταιριών αυτών και επίσης το αν συμμορφώνται εταιρείε του εταιρικού ευρωπαϊκού δικαίου. Πολλές φορές έχουμε κάποιες ειδικέ περιστάσεις που επιβάλλουν εξαιρετικού χαρακτήρα μέτρα, όμως να μην ξεχνούμε ότι κοστίζουν οι κρατικές ενισχύσεις, Στρεβλώντα ανταγωνισμό, οδηγούν σε ελλείμματα και χρέος κάτι το οποίο θα το κληροδοτούμε στις επόμενες γενιές. Άρα, συνάδελφοι, είναι καθήκον μας να δικαιολογείται και η τελευταία δεκάρα που ξοδεύεται. Οπότε η Οικονομική Επιτροπή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει και να αξιολογήσει ενδελεχώς ε, όλες αυτές τις ε, κινήσεις, το τι έχει γίνει δηλαδή όσον αφορά την Green Recovery και τις κρατικές ενισχύσεις πριν από δύο χρόνια είπαμε ότι δεχόμαστε αυτό το, αυτό το πακέτο μέτρων και την κρατική ενίσχυση ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια στροφή προς μια οικονομία βιώσιμης γνώσης. Έπιασαν το από τα λεφτά ρωτάμε σήμερα. Πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι ήταν οι επιλέξιμοι, τι κάνανε αυτοί όσον αφορά να έχουμε αυτή την ε, πράσινη ανάκτηση ας πούμε. Επομένως, να κάτσουμε να ρωτήσουμε αυτές οι κρατικέ ενισχύσεις τι στρεβλωτικά αποτελέσματα επέφεραν. Τώρα, όσον αφορά τις, ε, τις κάθετες συμφωνίες, η σχετική συμφωνία θα αναφερθεί φέτος. Έχει εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία Όμω, όμως απογοήτευσή μου κοίταξα και τελικά σε εφημερίδες βρήκα την τελευταία εκδοχή του κειμένου. Και όταν απευθύνω στην Κομισιόν και ρώτησα τι έγινε, πώς έγινε αυτή η διαρροή, τελικά εγώ δυσκολεύτηκα περισσότερο να τα βρω από τον τύπο. Άρα θα πρέπει να σταματήσει η Κομισιόν αυτές τις διαρροές προς τα ΜΜΕ. Και όταν αρνούνται τις διαρροές, αυτό προσβάλλει την νομοσύνη μας. Για την ουσία τώρα, ναι, ναι πρόεδρε, τελειώνω. Επί της ουσίας αυτής, οι πρώτες Ευρωπαϊκές επιτροπής ο, οδηγούν σε θεσμενή διάκριση κατά Αυτόν που ασχολούνται με το λιανεμπόριο σε σχέση με το One Stop Shop το 21ο αιώνα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό όχι να φημώνουμε, όχι να εμποδίζουμε τους online retailers άρα θα πρέπει όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν εδώ και πολύ καιρό να τα κάνει η Κομισιόν κυρίως όσον αφορά τις διαφημίσεις του Ιντερνετ και αν δεν θέλει η Κομισιόν να κάνει αυτό το περιστούμε, ας μας δικαιολογήσει το γιατί. Τέλος. Επίτροπε, έξι λεπτά μου είπατε. Έξι μου είπατε. Όχι, όχι, όχι, υπάρχει παρεξήγηση. Τέσσερα, τέσσερα λεπτά είπαμε, λέει ο πρόεδρος. Δεν πειράζει, τελειώστε όμως. Σχεδόν τέλειωσα, πρόεδρε. Επίτροπε, χαιρετίζουμε τη δέσμευση του Επιτρόπου Αλμούνια να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη διαμόρφωση τη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Γιατί η οικονομική κρίση κατέδειξε ότι χρειάζεται να έχει η πολιτική ανταγωνισμού μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα. Επομένω, μάλλον λάθο ήταν αυτό το οποίο έγινε με το έγγραφο που δεν πήραμε και πήγε στον τύπο. Άρα και για τη συνέχεια αυτής της διαδρομής ελπίζουμε να συνεργαστεί στενά μαζί μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε πώς και πώς την ε, απάντησή της. Ε, Πέντε λεπτά. Ο κύριος Μπαρνιέ, της Επιτροπής. Euh, Θα ήθελα και εξ ονόματος του, ε, του συναδέλφου και φίλου Χωακή Μαλμούνια να ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Ιντεβέλτ και βεβαίω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις ε, εισηγητέ από τι δύο αντίστοιχε επιτροπέ, ε, συνεισέφεραν και εκείνοι σε την προετοιμασία του, της έκθεσης αυτής. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου αναφέρεται σε πάρα πολλά θέματα, τα ακούσαμε μάλιστα, πολιτική ανταγωνισμού καθώς επίσης ε, και αναθεώρηση ε, του κανονισμού για τις ε, συγκεντρώσεις. Θεωρούμε ότι με την πολιτική ανταγωνισμού, την νέα έκθεση παίρνουμε καινούρια ε, βήματα για τον ανταγωνισμό και θα δώσει και τη δυνατότητα η έκθεση αυτή ε, να ξεκινήσει ένας ε, πολύ καλός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε ξεκινήσει και με τον κύριο Αλμούνια. Βεβαίως ο διάλογος αυτός ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει μια σωστή πολιτική σχέση και βεβαίως στα πλαίσια της συναπόφασης τα πράγματα γίνονται ε, ακόμα πιο ε, σαφή. Ε, βεβαίω δεν μπορεί να αλλάξει η νομική βάση της πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά μπορούμε να δούμε εάν αναπερίπτωση μπορεί η συναπόφαση να εφαρμοστεί σε επιμέρους αποφάσεις της πολιτικής ανταγωνισμού. Επ' αυτού γνωρίζετε ότι το προηγούμενο Ιανουάριο ο Επίτροπος Αλμούνια είχε ε, ανακοινώσει ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω θα συμμετάσχει ενεργά στην αντιμετώπιση του θέματος των προσφυγών ε, των ε, μεμονωμένων ε, ενδιαφερομένων. Βεβαίω, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και όσον αφορά το θέμα των συγκεντρώσεων δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολιτική διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα και βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού κυρίως σε μια τέτοια περίοδο κρίσης. Το 2008 ξεκίνησε η οικονομική οικονομική και χρηματοπιστωτική ε, κρίση και ε, ε, βεβαίως ε, ε, η τότε έκθεσή μας για την πολιτική ανταγωνισμού κατάφερε να ξεπεράσει μέχρι ένα μεγάλο βαθμό τα προβλήματα της κρίσης του 8. Όσον αφορά τώρα για το 2009 βεβαίως η μεγαλύτερη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στο ξεπέρασμα της κρίσης η οποία έχει βαθύνει ευθύνη το, το 2009. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επικοδομητικό διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ε, κυρία ε, Ιντεβέλτ, αναφερθήκατε επίσης στο θέμα ε, των εγκάρσιων των κάθετων περιορισμών. Θεωρούμε ότι έχει βρει η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μια ισορροπία αφενός ε, βάση των ε, προτάσεων για συνένεση μεταξύ των εμπορευομένων και πράγμα που τους επιτρέπει να βρουν τον καλύτερο τρόπο να προωθήσουν το προϊόν τους και βεβαίως να προστατεύσουν την εικόνα της μάρκας τους και ε, τους δίνεται πλέον η δυνατότητα ε, να προωθήσουν τις ε, πωλήσει τους σε φυσικά σημεία πώληση. Επίσης όσον αφορά το λιανεμπόριο online είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριτή αναφέρθηκε στα καρτέλ. Τα καρτέλ υπάρχουν και γνωρίζω ότι στην Ιρλανδία ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργίας πολλοί αγρότες πιστεύουν ότι δημιουργούνται τα καρτέλ διότι σιγά σιγά γίνονται όλο και πιο δύσκολη η επιβολή ρυθμίσεων και τα μεγάλα εργοστάσια είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τα κατέλη με τις μεταφορές των ζωζών κατά τρόπο που τους βολεύει και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών τα οποία ε, κοστίζει ο τομέας ε, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διαφορά μπορεί να είναι από 50 μέχρι 200. Και γι' αυτό νομίζω θα ήταν καλή πρωτοβουλία ε, να ελεγχθεί αυτό ο τομέας και να ληφθεί κατάλληλη δράση. Ευχαριστώ. Ο ε, κύριε Πρόεδρε, δεν σας ρώτησα πόσο χρόνο μου δίνετε. Φαντάζομαι ένα λεπτό. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίαση και θα ήθελα να πω ότι ο έλεγχο ε, των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού κυρίως γίνεται προ όφελο του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό και για τις επιπτώσεις για τον καταναλωτή η δύσκολη φάση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου περί ανταγωνισμού, ιδίως για τα θέματα των ενισχύσεων και των κρατικών ενισχύσεων, θα μας απασχολήσει. Δεν φαίνεται να υπήρξε πρόβλημα το 2008 και θα πρέπει η Επιτροπή κατά τον έλεγχο να φροντίζει η ευρωπαϊκή Ενία αγορά και οι ευρωπαίοι καταναλωτές να μην πλήττονται πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος που θα αφιερωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί θα πρέπει ε, να φροντίζουμε μέσω του δικαίου του ανταγωνισμού να μην πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. αυτό το οποίο ε, προτείνεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να αποδεχθούμε. για ένα λεπτό. Το 2008 άνοιξε το κεφάλαιο για το τι κάνουν τα καρτέλ τους καταναλωτές και επομένως είπαμε ότι θέλουμε να έχουμε όλα αυτά τα κατασταλτικά πρόστιμα, να έχουμε τις συνοδευτικές οδηγίες, ε, την Λευκή Βίβλο για να μπορέσουμε να βάλουμε μια ευταξία στον ανταγωνισμό μέσα σε αυτή την ε, συγκυρία της κρίσης οι κρατικές ενισχύσει κάπως αντιστάθμισαν ε, τις ζημιές και θα πρέπει όμως να μην έχουμε τον κίνδυνο της στρέβλωσης προσοχή όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, της ΜΜΕ, τη διατροφική αλυσίδα και θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία του τι γίνεται με τα γαλακτοκομικά και χρειάζεται επομένω να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό το αποτέλεσμα τη έκθεση και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Το. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ήμουν ε, σκιοδησηγητής, οπότε πρώτα-πρώτα θέλω να συγχαρώ την συνάδελφο Σόφι Νετφέλτ, διότι ε, νομίζω ότι εξεπώνησε μια πάρα πολύ ποιοτική έκθεση. Νομίζουμε ότι θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το θέμα που αφορά τι κρατικέ ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την οικονομική κρίση. Έγινε δυνατόν να επιτραπεί στα κρατημέλη να παράσχουν τέτοιε ενισχύσει υπό κάποιε προποθέσει σε κάποιε εταιρείε, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάτσει και να ελέγξει κατά πόσον αυτέ οι ενισχύσει ε, χορηγήθηκαν με τρόπο σύνομο και ποια ήταν τα αποτελέσματα. Διότι θέλουμε να μην έχουμε στρέβλωση στην ε, αγορά και να μην παροξενθεί η κακή οικονομική κατάσταση. Ούτε να πληγεί όλος ο κόσμος από αυτή την οικονομική κρίση. Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ανταγωνιστική ε, ενεργειακή αγορά και έτσι επομένω να φροντίσουμε την νέα αγορά. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαρθεί αυριο αύριο, 3η 9 Μαρτίου 2010, από 9 με 1 3 με 7.30 και 9 με 12 τα μεσάνυχτα. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έληξε. Καληνύχτα σε όλους σας αγαπητοί συνάδελφοι.